μέλη με βάση τον κανόνα της ενισχυμένης συνεργασίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για αυτό το θέμα ε, της τη ημερήσια διάταξη. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι στι 12.30. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα λοιπόν ε, που είναι η έκθεση του κυρίου Βοητσεχόφσκι για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Άρχεται η συζήτηση, θα δώσουμε στο λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ απαράδεκτο στην Ευρώπη του 21ου αιώνα να δείχνουμε αναισθησία ή απαθροπιά απέναντι στα ζώα. Γιατί και τα ζώα είναι ζωντανά πλάσματα, πολύ ευαίσθητα, που αισθάνονται τον πόνο, την οδύνη. Δεν θα πρέπει να τα βασανίζουμε λοιπόν. Και θέλουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στη μεταφορά των ζώων και αυτό ασχολούμαστε με την έκθεση αυτή. Λάβαμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταφορά των ζώων, των ζωντανών ζώων, που είναι όλο και περισσότεροι, 30 εκατομμύρια ε, ε, ε, γουρούνια, 8 εκατομμύρια βοηδοί. έχουμε 2 τρίτα των ε, μεταφορών αυτών που διαρκούν πάνω από 8 ώρες. Και με εξαίρεση τη μεταφορά των αλόγων αυξάνονται οι μεταφορές των υπόλοιπων ε, ζώων που για μεγάλο διάστημα μεταφέρονται σε μακρινέ αποστάσει. Το ταξίδι κρατάει πάνω από 24 ώρε πολλέ φορέ και είναι δύσκολο να ελέγξουμε τέτοιου είδου μεταφορέ. Μάλιστα, ορίμασε η κατάσταση ώστε να πρέπει να συζητήσουμε πια σοβαρά την πρόταση πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων και ε, τον, την πρωτοβουλία των πολιτών που ζητούν να περιοριστεί το πολύ σε οκτάωρο η μεταφορά των ζωντανών ζώων. Και χαίρομαι που στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου η έκθεση πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία. Πολύ συντομότερες μεταφορές ε, είναι καλύτερες για τα ζώα και για τους καταναλωτές γιατί έτσι αποφεύγουν ε, το πολύ στρες στα ζώα και έτσι ε, δεν δημιουργούνται τοξίνες στο σώμα τους. Επίσης, οι σύντομες μεταφορές είναι λιγότερο δαπανηρές, γιατί οι μεταφορές μεγάλης αποστάσεως είναι πολύ πιο δαπανηρές ε, και έτσι χάνουν και οι κτηνοτρόφοι και ταυτόχρονα οι καταναλωτές που αναλαμβάνουν ακόστος των μεταφορών καλούνται να πληρώσουν περισσότερο για το κρέας που αγοράζουν. Οπότε με συντομότερες μεταφορές θα έχουμε λιγότερες οδικές μεταφορές, λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, περισσότερη τοπική παραγωγή, εκτροφία κοντά στους ε, πολίτες, παραγωγή κοντά στην κατανάλωση. Όλα αυτά είναι θετικά για όλες τις πλευρές. Στην πρότασή μου προτείνονται πολύ σημαντικές προτάσεις προκειμένου να περιοριστούν σε οκτάωρο οι μεταφορές ζωντανών ζώων. Είναι πολύ σημαντικό το μέτρο. Δεν λέμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ε, χωρί καμία εξαίρεση. Λαμβάνονται υπόψη κάποιε γεωγραφικέ ιδιαιτερότητε, τα νησιά ή εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Θέλουμε με την έκθεση αυτή να συνεχίσουμε τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να κοφεύουμε απέναντι σε κλήσει των συμπολιτών μα, γιατί πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν αυτή την πρωτοβουλία για περιορισμό της μεταφοράς ζωντανών ζώων σε οκτάωρο το πολύ. Δεν μπορούμε να μακοφεύουμε και να εθελοτυφλούμε μπροστά σε τέτοιες ε, ε, κλήσεις. Δεν θα πρέπει ε, να με εμένει πεισματικά σε όχι και να μην προτείνει μέτρη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε σε τόσο προχωρημένο πολιτισμό να δείχνουμε αναισθησία απέναντι στα ζώα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ενέκριναν χωρίς τροπολογίες την έκθεση και πιστεύω ότι χάρη στην εργασία και στη Γεωργική Επιτροπή καταλήξαμε σε πολύ λογική και συνετή λύση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας αλλά και ε, τα μέλη της ομάδας για την ευζοία, για την αμέριστη και καρποφόρα συνεργασία που είχαμε. Στα αγγλικά. Κυρίες και κύριοι, ο Μαχατ Μακάντι είπε ότι το μεγαλείο ενός λαού ε, και η πρόοδος του η ηθική κρίνεται από, το από τον τρόπο που μεταχειρίζεται τα ζώα του. Οπότε τα ζώα που καταναλώνουμε ε, στην οικονομία μας και ο τρόπος που τα μεταχειριζόμαστε μάλλον δεν θα αλλάξει στο εγγύς Αλλά ε, ήδη από τώρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τις οδύνες, τα βάσανα αυτών των ζώων κατά τη μεταφορά. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι δυνατόν να μειώσουμε τα βάσανά τους ε, όπου γίνονται τις μεταφορές και όπου χρησιμοποιούμε αυτά τα ζώα. Ο περιορισμός του χρόνου μεταφοράς είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και υπάρχουν ήδη επιστημονικά πορίσματα ε, που συνάδουν προς κάτι τέτοιο και θα είναι απόδειξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού του 21ου αιώνα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος, κύριος Μπόρκ, παρακαλώ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία σήμερα να μιλήσω στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα που είναι και ευαίσθητο και συναισθηματικά φορτισμένο και αφορά και ενδιαφέρει τόσο πολλούς βουλευτές και εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Βεβαίως, υπάρχει διάσταση απόψεων για τη μεταφορά των ζώων και το ανώτατο όριο της διάρκειας. Βεβαίως θα πρέπει πάντα να εφαρμόζονται τα σωστά πρότυπα το Νοέμβριο του 2011 ενέκρινε πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταφορά των ζώων και αυτό ε, σύμφων, σήμαινε ε, εφαρμογή του κανονισμού 2005 αριθμών 1 ε, θα πρέπει όμως να βελτιωθεί και έπρεπε να έχει βελτιωθεί η κατάσταση δεν εφαρμόζεται ακόμα επαρκώς ο κανονισμός ο ισχύων και η κείμενη νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστότερα έρχομαι τώρα ε, στο μεγάλο έργο της έκθεσης του εισηγητού κ. Βουτσικόφσκη και τον ευχαριστώ και είμαι ευγνώμων για τις προσπάθειές του για την περίπλοκη αυτή υπόθεση. Ένα από τα πιο επίμαχα θέματα είναι ανώτατη διάρκεια της μεταφοράς και ένα από τα συμπεράσματα ε, που μπορούμε να βγάλουμε από τη δότηση πρόσφαση της ΕΦΣΑ είναι ότι δεν υπάρχει επιστημονική δικαιολογία για να υπάρχει όριο 8 ώρων ε, για όλα τα είδη ζώων και υπό όλες τις συνθήκες. Θα πρέπει να να λαμβάνουμε υπόψη όλες ε, τις συνθήκες και όλες τις πτυχές μεταφοράς. Χαίρομαι που η έκθεση υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάγκη να βελτιωθεί η εφαρμογή γιατί ε, και, όλες αυτές, ε, και πολλές από τις προτάσεις έχουν γίνει και από εμά. Εναρμόνιση ε, τον τρόπο με τον οποίο αναφέρουν τους ελέγχους στα κράτη-μέλη και έχω τη χαρά κύριε Πρόεδρε σήμερα να σας ανακοινώσω ότι η σχετική εφαρμοστική πρόταση το σχέδιό της θα συζητηθεί με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχάς του επομένου έτου Επίσης να αναφέρω δύο από τις δραστηριότητες ε, του ΕΦΙΟ e που είναι η υπηρεσία τροφίμων και κτηνιατρική ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα κράτη-μέλη για να ανταλλάσσουν ευέλτιστες πρακτικές σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού 1 κάθετος 2005 και το 2013 μια νέα σειρά επιτόπου επισκέψεων ε, θα ενισχύσουν τις προσπάθειές μας και θα έχουμε έναν επιθεωρητή ε, του Γραφείου ε, Τροφίμων και κτηνιατρικών υποθέσεων και ε, εμπειρογνώμονε από μια χώρα που θα επισκέπτονται άλλε χώρε. Για του εξή δύο λόγου θα γίνονται αυτέ οι επισκέψει. Θα έρχονται υπάλληλοι ε, των κρατών μελών με ιδιαίτερα προβλήματα σε άλλα κράτη ε, που εφαρμόζονται καλύτερα και αντιμετωπίζονται οι καταστάσει. Και επίση οι επιθεωρητέ θα πηγαίνουν προς τους ε, ίδιους εμπορικούς δρόμους που ακολουθούν και οι μεταφορές των ζώων. Ας πούμε από την Ολλανδία θα πηγαίνουν στη Γερμανία, στην Ιταλία, όπου γίνεται όλο το δρομολόγιο της μεταφοράς χείρων επί παραδείγματι. Ε, υπάρχουν και άλλες ε, πρωτοβουλίες που ετοιμάζουμε. Ε, βελτίωση των ελέγχων στη μεταφορά των ζώων με καλύτερη χρήση των συστημάτων πλοήγησης τρόποι ερμηνείας των κανονισμών, διεθνή συνεργασία για ενίσχυση της ευημερίας των ζώων σε τρίτες χώρες και επικοινωνία και ανακοινώσεις προς τους πολίτες. Επίσης συνεργαζόμαστε με τον κλάδο και ΜΚΟ για να προωθήσουμε ε, και ε, πρωτοβουλίες για ενημέρωση. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις όμως στην έκθεση με τις οποίες δεν μπορεί να συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά αυτό το μεγάλο αριθμό περίπλοκων μελετών και ε, εκθέσεων που ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να κάνει εκθέσεις όταν πρόκειται για ειδική πρωτοβουλία. Επίσης, δεν συμφωνώ με την άποψη ότι η κείμενη νομοθεσία για την υγιεινή και την ευημερία των ζώων ευθύνεται ε, αμέσω για την αύξηση της διάρκειας και ε, της μεγάλης αποστάσης που μεταφέρονται τα ζώα. Επιτρέπουμε ε, ε, να παραμένουν τα μικρά σφαγεία οικονομικά βιώσιμα αλλά θα πρέπει να σέβονται τις συνθήκες υγιεινής και ευημερίας. Ε, τέλος θα ήθελα να πω ότι εκτιμούμε πολύ το ενδιαφέρον και την προσήλωση του Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα. Ακόμα και αν διαφωνούμε με κάποιες λεπτομέρειες, γενικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κοινό στόχο να βεβαιωθούμε ότι τα ζώα θα μεταφέρονται με τρόπο που θα επιτρέπει την ευημερία τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πίτροπε, περνάμε τώρα στις ε, γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών. Έχουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος ε, Υγείας ε, και Ασφάλεια Τροφίμων που μας την, θα μας την παρουσιάσει η κυρία Μαρτίνα Άντερσον. Παρά την, τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη μεταφορά των ζώων που υπάρχει από το 2005, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Ο κανονισμός δεν έχει εφαρμοστεί, κυρίως λόγω του ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με αυτόν. Πρέπει λοιπόν ε, να αντισταθούμε σε περιτά ταξίδια των ζώων για σφαγή. Ε, παραβιάζονται τα κριτήρια της καλής διαβίωσης ε, των ζώων. Τα μακρινά ταξίδια ενέχουν τον κίνδυνο κακής υγιεινής και ως εκ τούτου της μετάδοσης και διάδοσης ασθενειών. Εκτός αυτού τα ζώα που είναι κάτω από στρες παράγουν τοξίνες που επηρεάζουν την ποιότητα του να έχουμε λοιπόν μικρές αποστάσεις. Μέχρι 6 εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται ζώα ε, για σφαγή ε, κάθε χρόνο. Είναι ε, ένα ζωικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να λαμβάνουμε πλήρως υπόψη μας και να το σεβόμαστε. Ευχαριστούμε εκ μέρους της Επιτροπής Μεταφορών ο συνάδελφος κ. Ντεγκράντες Πασκουάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διάρκεια τη μεταφοράς είναι μία επιπλέον παράμετρος που επηρεάζει την ευζοία. Δεν έχει νόημα ή δεν εξυπηρετεί τίποτα να περιορίσουμε σε 8 ώρες τη μεταφορά αν δεν είναι εξοπλισμένα κατάλληλα τα οχήματα ώστε να έχουν κατάλληλο εξαερισμό ε, και να έχουν οι μεταφορεί οδηγοί την κατάλληλη κατάρτιση για να ξέρουν να μεταχειρίζονται ζώα. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και η κοινοτική νομοθεσία είναι από τις πιο φιλόδοξες του κόσμου. Οι επιστήμονες της ε, ε, Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων ε, λέει ότι η ευημερία των ζώων εξαρτάται περισσότερο από τις συνθήκες μεταφοράς και όχι τόσο από τη διάρκεια. Είναι ισορροπημένη η έκθεση και έλαβε υπόψη τη γνωμοδότηση τη Επιτροπής Μεταφορών. Όλες αυτές οι διακηρύξεις και τα λόγια είναι πολύ ωραία, αλλά και φυσικά έχουν ένα τμήμα τη αλήθεια, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Τα συμφέροντα των χωρών που ενδιαφέρονται να εξαγάγουν ε, κατεψυγμένα ζώα. Γιατί δεν του ενδιαφέρει η μεταφορά ζώων των ζώων. Γιατί δεν εφαρμόζουμε τι ίδιε διατάξει και για τα ζώα που, ε, για τα ζώα που μεταφέρονται προς πάχηση και όχι απλώ προς φαγή, λόγω των συμφερόντων που κρύβονται πίσω από τι προτάσει. Ευχαριστώ. Εξ των πολιτικών ομάδων. Τώρα πρώτη η κυρία Στέρντε από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπόθηκε ήδη ότι για το ΕΛΚ η νομοθεσία για τη μεταφορά των ζώων είναι σημαντικό και στον ιδανικό κόσμο ε, βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και ε, είναι πολύ σημαντική και η διάρκεια ε, για την ευημερία. Αλλά ξέρουμε ότι ο πραγματικός κόσμος πόρο απέχει από τον ιδεώδη. Ε, το 2004 έκανε μια πρόταση ε, το Συμβούλιο για τις συνθήκες μεταφοράς. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και πραγματικά να τιμωρούνται εκείνοι που ε, σφάλουν και δεν εφαρμόζουν σωστά. Είναι χίλιος πτέρνα και πάλι θα πρέπει να ξαναγίνει στο νέο κανονισμό αυτό το θέμα του ελέγχου και των επιθερήσεων. Να μην είναι τα σχήρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ότι δεν την αφορά και αρμόδια είναι τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το προσέξει. Γιατί αγαπητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεστε να διαπιστώνετε ότι υπάρχουν διαφορές στους ελέγχους και μεγάλες μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά δεν κάνατε ε, ε, περισσότερες επιθεωρήσεις του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων το περασμένο χρόνο. Και είναι και διαφορετικές οι όταν αφορά ε, την ε, μεταφορά των εμπορευμάτων το κάνετε, αλλά όταν πρόκειται για ζωντανά πλάσματα, για ζώα δεν το πράτετε. Κατά την άποψή μου αυξάνεται η πίεση και καλά κάνει και θα πρέπει να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα της μέγιστης διάρκειας. Αύριο θα ψηφίσουμε την πρόταση του εισηγητή για το οκτάωρο. Και αύριο πραγματικά θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ψηφοφορία. Ε, την τελευταία φορά που κάναμε αυτή την πρόταση δεν είχαμε συναπόφαση. Τώρα έχουμε. Γιατί άραγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει φέρει ε, πρωτοβουλία νομοθετική για αυτό το θέμα. Δεν μπορείτε να κρύβεστε πίσω από μια συμφωνιούλα με το Συμβούλιο. Αύριο θα ε, ψηφίσουμε και θα πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία για το ψήφισμα για τη μέγιστη διάρκεια 8 ώρων στις μεταφορές. Υποστηρίζουμε πλήρως τον εισηγητή. Ευχαριστώ η κυρία Κάντενμπαχ. Αξιότιμε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, από το 1997 σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν διατάξεις για την ε, προστασία των ζώων. Αυτές έτυχαν επεξεργασία το 2005 και τώρα ε, έχει καταδειχθεί ότι υπάρχουν βελτιώσεις ε, αλλά δεν είμαστε παρόλα αυτά ικανοποιημένοι. Ε, δεν θέλω να συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπε η προλαλήσασα διότι κύριε Επίτροπε θέλουμε να σας δώσουμε την ευκαιρία να μετρηθείτε με το παρόν και το μέλλον και όχι με το παρελθόν. Εμείς λοιπόν επιθυμούμε να υπάρχει μια νομοθεσία που θα εγγυάται ότι ε, ισχύει η προστασία των ζώων και μία από τις προτάσεις που έχουμε είναι να τηρείται το οκτάωρο και αυτό ε, εφόσον υπάρχουν ε, επιστημονικά τεκμηριωμένα ε, στοιχεία. Υπάρχει ένα εκατομμύριο Ευρωπαίων που τάχθηκε υπέρ του οκτάωρου. Έχουμε τη γραπτή σχετική δήλωση που εγκρίθηκε και υπογράφηκε και από εμάς. Ο κανονισμός αυτός ε, δεν ξέρουμε αν μπορεί να εφαρμοστεί. Πρέπει να υπάρχει ένας άλλος κανισμός, ο οποίος ε, θα επιτρέπει τον έλεγχο. Από την άλλη όμως ε, οι περιοχές που δεν μπορούν να τηρήσουν το οκτάωρο να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες όμως δεν πρέπει να συμβάλλουν στην αποδυνάμωση του κανονισμού. Εμείς επιθυμούμε ε, να μειωθεί ο αριθμός των ζώων που μεταφέρονται στην Ευρώπη. Επιθυμούμε να περιοριστεί ο αριθμός των μεταφορών και επιθυμούμε να περιοριστεί η διάρκεια των ταξιδιών. Αυτό θα το πετύχουμε μόνο εφόσον υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι και εφόσον από τα κράτη-μέλη προσφέρονται στοιχεία τα οποία να είναι αξιόπιστα. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας δεν υπάρχουν οι απαραίτητες εγγύησεις. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, κύριε Επίτροπε να επηρεάσετε τα κράτη-μέλη και να μεριμνήσετε έτσι ώστε οι έλεγχοι που προβλέπονται στην έκθεση να εφαρμόζονται γιατί μόνο έτσι θα υπάρχει ουσιαστική προστασία των ζώων στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πόλσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας τον κύριο Βατζοχόφσκι για την έκθεσή του. Ε, είναι πολύ αξιόλογο το έργο σας και δείξατε μεγάλη υπομονή. Γνωρίζω τα θέματα προστασία των ζώων και ιδιαίτερα η ευζωία τους κατά τη μεταφορά. Είναι ένα θέμα που ε, ταράζει πολύ κόσμο και ενοχλεί πολλού. Μερικοί είναι υπερβολικά φιλόδοξοι, αλλά δυστυχώ, ε, στο περιβάλλον που ζούμε σήμερα, ε, κυρίως στο αστικό, έχουμε τόσο πολύ κόσμο που στερείται ειδικών γνώσεων για το φυσικό περιβάλλον που είμαστε υποχρεωμένοι μερικές φορές στις ε, αποφάσεις που λαμβάνουμε να κάνουμε συμβιβασμούς. Και οι συμβιβασμοί θα πρέπει να στηρίζονται στις πρόσφατες ε, επιστημονικές μελέτες και στα ε, τελευταία επιστημονικά πορίσματα. Από εκεί θα πρέπει να χαράξουμε την πορεία μας. Και τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για να λάβουμε τις αποφάσεις μας είναι σημαντικά. Μια δημοκρατική απόφαση όμως θα πρέπει να στηρίζεται και σε κάποια ε, κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, δεοντολογικά που θα συνοδεύουν τα επιστημονικά απορίσματα και τα επιστημονικά στοιχεία. Η Άλντε υποστηρίζει ολόψυχα την έκθεση του εισηγητού. Ένα αρνητικό μόνο πρόσημο έχουμε για την παράγραφο 14, εδάφιο 5. Εκεί βάλαμε αρνητικό πρόσημο στον κατάλογο ψηφοφορία, αλλά είναι το μόνο αρνητικό σημείο. Στα υπόλοιπα συμφωνούμε με τον εισηγητή. Ο κύριο Έκχοτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινέστατα τον εισηγητή ε, για να καταλήξουμε στην έκθεσή του και στην απόφαση. Και ε, για ε, την ευημερία των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Συμφωνώ απολύτως με το ψήφισμα όπως έχει σήμερα και όπως θα ψηφίσουμε. Νωρίτερα, ε, ή μάλλον το πω ε, είπαμε ότι υποστηρίζουμε το 8ωρο, αλλά η πρώτη εκδοχή του κειμένου δεν ήταν η σωστή. Στην αρχή ε, λέει ότι δεν είναι επιστημονικό και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ε, Επίτροπο να το εξετάξει, να κοιτάξει κάτι για το 8 κτλ. Αυτό παρά είναι ε, αδύναμο. Έχω φτιάξει ένα δικό μου ψήφισμα εναλλακτικό. Συμφωνώ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τον εισηγητή, εκτός όμως από αυτές τις δύο παραγράφους. Ε, και τις έχω αντικαταστήσει απλούστατα με την άμεση έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελάτε με νομοθετική πρόταση ε, που να ορίζει ανώτατη διάρκεια 8 ώρες με ε, τη δήλωση που έχει υπογράψει η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και εκατομμύρια πολιτών ζήτησαν. Συμφωνώ απολύτως με την έκθεση αλλά το 8 ώρο θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ε, μια ανυποχώρητη απέτηση του Κοινοβουλίου. Και κατά τα το ψήφισμα είναι καλό. Ευχαριστώ ο κύριος Τζέιμς Νίκολσον. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί την πάρα πολύ καλή δουλειά, δύσκολη δουλειά. Ε, ξέρουμε όλοι και το συναισθηματικό στοιχείο, το ανέφερε και ο Επίτροπος. είναι ένα φορτικά, συναισθηματικά φορτισμένο θέμα για πολλούς ανθρώπους τίθενται σημαντικά ερωτήματα και νομίζω ότι κανείς δεν είναι υπέρ της ε, περιττής μεταφοράς ζώων σε μεγάλες αποστάσεις. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες που να διασφαλίζουν ότι η μεταφορά είναι όσο πιο ανθρώπινη γίνεται. Είμαι ακράτα πεπισμένος ότι ε, πρέπει να εξάγουμε ε, τα προϊόντα του κρέατος, ε, να υπάρχουν ε, κινητά σφαγεία στην Ευρώπη. Εφόσον υπάρχουν αυτά, μπορούν να γίνονται μεταφορές και σε απομακρυσμένες περιοχές. Άρα είναι, υπάρχει πρόβλημα εδώ και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην καλή διαβίωση των ζώων, αποτελεσματικούς κανόνες και κυρίως εφαρμόσιμους κανόνες Όσον αφορά επίσης το θέμα αυτό, θα πρέπει αυτοί ε, να, λαμβάνονται υπόψη, να λαμβάνονται υπόψη και οι απομακρυσμένες περιοχές, να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση εις βάρος κάποιων περιοχών ή κρατών μελών και σίγουρα να μην υπάρχει και στρέβλωση του ανταγωνισμού. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος κύριος Ρούμπιτς. Ευχαριστώ. Θα Πιστεύω ότι ε, θα υποστηρίξουμε το ψήφισμα, αλλά τελικά τι επιθυμούμε. Εμείς ε, επιθυμούμε καταρχήν να υπάρχουν ε, μικρά σφαγεία που να υποστηρίζονται, να υπάρχουν, αυτό είναι και μέτρο κατά της ανεργίας. Κατά δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει ε, τη θερμοκρασία που πρέπει να επικρατεί κατά τη μεταφορά των ζώων, να υπάρχουν ποτίστρες και όλα αυτά ε, να είναι δεσμευτικά για τους ε, μεταφορείς. Να υπάρχει και εξαρισμός. Ευχαριστώ κυρία Τότς. excuse me. Α, συγγνώμη, ξέχασα τον κύριο Άγνιο προηγουμένω. Βιάστηκα. Μα πρόεδρε, έχουμε ήδη κατάλληλη νομοθεσία για την ευημερία των ζώων. Αυτό που λείπει είναι να εφαρμόζονται οι κείμενοι κανόνες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε δύο φορεί που επιθεωρούν και συχνά βρίσκονται σε σφαγεία, σε ε, κρεαταγορές όπου φορτώνονται τα ζώα και εξεφορτώνουν. Και Επίσης, ε, ε, κοιτάνε τις προδιαγραφές, αν υπάρχει σωστός κλιματισμός, εξαερισμός, πώς είναι τα κλουβιά, ε, αν είναι ίδιες οι διαστάσεις, αν έχει προβατίνες έγκυες, τα διάφορα είδη των ζώων μεταφέρονται μαζί, αν γεννούν σωστά τα ζώα και οι άνθρωποι διώκονται όταν δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία. Δεν μου αρέσει ε, να μας λένε ε, πώς ε, θα μεταφέρουμε τα ζώα μας κάποιοι άνθρωποι που διοργανώνουν τα βρομαχίες και άλλα τέτοια. Αυτά είναι πολιτική και ιδεολογία και τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ. Τώρα με τη σωστή σειρά θα δώσω το λόγο στην κυρία thank Τότς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή μα για το έργο του στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Είναι όντω συναισθηματικό θέμα, συγκινησιακά φορτισμένο. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αλλοιωθεί, να εξουδετερωθεί την καλή προσπάθεια που έκανε η Επιτροπή Γεωργία και γενικώ ε, ο γεωργικό κλάδο. Χρειαζόμαστε προδιαγραφέ για να βελτιώσουμε τη διαβίωση των ζώων στι μεταφορέ. Ε, καλύτερη κατάρτιση ε, των μεταφορέων, ε, προβλέψεις για διακοπή και ανάπαυλα και κατάλληλο εξοπλισμό των οχημάτων. Όλα αυτά είναι σημαντικά στις μεταφορές. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ολόκληρο τον κλάδο να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές και να συμμορφωθεί με τις νομοθετικές διατάξεις. Όμως, όπως όμως και πολλές άλλες ε, κοινοτικέ προτάσεις, χρειαζόμαστε καλύτερη σαφήνεια για να αποφύγουμε την αβεβαιότητα και τις αφησιμίες. Έτσι θα αποφύγουμε τις παρερμηνίες των κανόνων και την διαφορετική εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κανονισμό που κατά τη γνώμη μου δεν εφαρμόζεται σωστά ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πριν εγκρίνουμε νέους κανονισμούς θα πρέπει να διορθώσουμε τη μη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό και επηρεάζει και τις ε, ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές γιατί μερικές φορές περιορίζει τις εξαγωγές των ζωντανών ζώων, εκθέτει τους γεωργούς ε, στη, στο έλεος των τοπικών σφαγίων που ε, δημιουργούν μονοπωλιακή και δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Χρειαζόμαστε υψηλέ προδιαγραφέ για την ευζοία, αλλά και σωστή ισορροπία μεταξύ του εύχριστου, του πρακτικού και του ε, εφαρμόσιμου νομοθετικά και στην πράξη. Ευχαριστώ κύριε Γέγκλε. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον εισηγητή μας Πραγματικά πολύ συναισθηματικά φορτισμένο το θέμα, αλλά έκανε καλή δουλειά. Και τελικά, κατά τη γνώμη μου, είναι καλό και το αποτέλεσμα. Και αν ψηφίσουμε αύριο όπως προτείνει. Περί τίνος πρόκειται εδώ. Είναι ζώα που προορίζονται για σφαγή, όχι για εκτροφή και πολύ λιγότερο κατοικίδια ζώα ε, που συνήθως ε, μεταφέρονται με τον καλύτερο τρόπο χρειάζεται έλεγχος εναρμονισμένος για την εφαρμογή των ισχυών των κανονισμών στα κράτη-μέλη. Είναι δηλωμένος μας στόχος να έχουμε ε, συγκρίσιμους ε, κανόνες με ίσο ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, αυτή η καλή ε, έκθεση δεν θα πρέπει να αναχθεί στο αν ε, περιλαμβάνεται ε, η μέγιστη διάρκεια των 8 ωρών. Αυτό είναι ένας ε, όρους ε, έτσι για να προσανατολίζεται κανείς και όχι απόλυτη προϋπόθεση. Υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες για τη φόρτωση, για την εκφόρτωση και για τη μεταφορά. Εγώ είμαι ευγνώμων για τα όσα επιτύχαμε και θέλω και πάλι να τονίσω ότι θα πρέπει να ε, δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και ε, στη μεταφορά αλλά και στις συνθήκες που ισχύουν, τις συνθήκες πλαίσιο και να είναι εγγυημένη η εφαρμογή του κανονισμού. Τρίτον, ο αριθμός των ζώων που μεταφέρονται στην Ευρώπη γενικά θα πρέπει να μειωθεί. Υπό την έννοια αυτή το Κοινοβούλιο απαιτεί σε αυτό ε, και σε αυτή την έκθεση αλλά και στο δεύτερο πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής μικρούς χρόνους μεταφοράς με τοπικά σφαγεία, μικρά σφαγεία και τελικά ε, να μεταφέρεται το κρέας ε, και όχι τα ζώα που προορίζονται για σφαγή. Θα είχε νόημα, υπήρχε, εμεί το καταστρέψαμε με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά και το κατεψυγμένο κρέας ε, που έρχεται ε, από μακριά και υπερατλαντικά το τρώνε. Οι ε, καταναλωτές θα μπορούσαν να ισχύει το ίδιο και για κρέας που προέρχεται από ζώα που σφάζονται κοντά στον τόπο κατανάλωση. Ο κύριος Αντρίου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ πολύ με τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής και με το ισορροπημένο έργο του εισηγητού μα Βοητσεχόφσκη και τον, τον οποίο και συγχαίρω. Η ισχύουσα νομοθεσία επέτρεψε την βελτίωση της κατάστασης ό,τι αφορά τη μεταφορά ζώων προς φαγή. Αλλά απομένουν πολλές προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να εφαρμόζονται ομοιόμορφα οι υπάρχοντες κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, να καταλήξουμε σε βέλτιστες πρακτικές και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ χωρών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι η νομοθεσία για τον περιορισμό της μέγιστης διάρκειας σε 8 ώρες που εξετάζεται ακόμη θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά λαμβάνοντας υπόψη κάποιες εξαιρέσεις όπως ε, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, την κατάσταση του οδικού δικτύου ή τις απρόβλεπτες καθυστερήσεις που είναι ανεξάρτητες ε, και εκφεύγουν του ελέγχου του μεταφορέα. Όπως είπε η Επιτροπή, ε, στη, με βάση την εφιστάμενη νομοθεσία δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις. Ο κύριος George Λάιον. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, πολύ συχνά το θέμα της μεταφοράς των ζώων γίνεται έρμεο του απλουστευμένου απλοϊκού επιχειρηματός ότι ο ότι οτιδήποτε κάτω των 8 ώρων είναι καλό για τα ζώα και ε, άνω των 8 ώρων είναι κακό για τα ζώα. Ασχολήθηκα με την εκτροτροφία πολλά χρόνια και σας διαβεβαιώ ότι ο περιορισμός στις 8 ώρες και το ρώσιμο αυτό είναι τελείως εσφαλμένο και δεν στηρίζεται και σε επιστημονικά πορίσματα. Και μάλιστα για τους χείρους και τα άλογα αναφέρεται ότι όντως θα πρέπει η μεταφορά να είναι συντομότερη. Για τα βοηδή όμως, ε, τα χοιρινά και τα πρόβατα το στρες δημιουργείται όχι μόνο, ε, όχι εξαιτία τη ε, παράταση του ταξιδιού άνω των 8 ώρων, αλλά από την ε, φόρτωση και εκφόρτωση των ζώων και τι μεταφορτώσει. Αυτό είναι που δημιουργούν περισσότερο το άγχο στα ζώα, το στρες και όχι η διάρκεια του ταξίδιου καθ' Θα πρέπει να ακούσουμε την Επιτροπή που λέει το πρόβλημα έγκυται στην ελληπή συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία. Αυτό είναι σκανδαλώδε. γιατί για τη μεταφορά των ζώων έχουμε πολλές διατάξεις, έχουμε περιορισμούς στις, ε, ε, στις προδιαγραφές ε, των κλοβών και πολύ ψηλέ προδιαγραφές για τον εξοπλισμό, αλλά δεν εφαρμόζονται. Το κλειδί για τη βελτίωση της ευζοίας είναι η εφαρμογή και η συμμόρφωση με την παρούσα νομοθεσία. Ε, σε ό,τι φορά τα τοπικά σφαγεία, συμφωνώ με την κυρία Γέγκλε. Θέλουμε όλοι πολύ περισσότερα μικρά τοπικά σφαγεία, να γίνουν αυτά πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι με τα τρακόντια μέτρα που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το ε, όνειρο να επαναφέρουμε τα μικρά τοπικά σφαγεία ποτέ δεν θα γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Το λόγο κύριος Καρλ Σλούτερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Από το 1995, από την ε, ένταξη της ε, Σουηδίας, περιμέναμε να υπάρξουν ε, μικρότερες διαδρομές, αλλά θέλουμε και καλύτερες συνθήκες κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής και καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας. Αυτός ο κανονισμός των οκτώ ωρών ε, διευκολύνει. Βεβαίως τα όρια δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Πολλά ζώα ε, δεν νιώθουν καλά όταν βρίσκονται σε άγνωστο περιβάλλον. Ε, το πιο δύσκολο είναι το πρώτο λεπτό στη μεταφορά. Το πόσο μπορούμε να δεχτούμε το χρονικό διάστημα της μεταφοράς, αυτό είναι και πολιτικό και ηθικό θέμα. Ε, γιατί εκλείονται ορμόνες ε, στρες. Επίσης ε, έχουμε περιμείνει αρκετό καιρό έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει μία πρόταση το συντομότερο δυνατόν που θα εξετάζει όλες τις πτυχές του θέματος, όχι μόνο τη μεταφορά. Ευχαριστώ κυρία Τζούλη Γκέρλινγκ. Thank you, Mr. President. I'd also like to... Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου κύριο Βοητσικόφσκι ε, για την ακάματη εργασία του και την υπομονή του. Θα ήθελα όμως να πω το εξής και αυτό συνδέεται με το εξής γεγονός. Το 2010 η πρώτη πρώτη γραπτή δήλωση που ήρθε στο Κοινοβούλιο και κυκλοφόρησε και η πλειοψηφία ε, καλούσε το Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κοιτάξει ε, την ιδιαίτερη περίπτωση των υποειδών που μεταφέρονται για σφαγή. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει έχουν πολύ τεκμηριωμένα στοιχεία για τη μεταφορά των αλόγων και ε, ο προκάτοχο του Επιτρόπου το έχει συζητήσει σε βάθο. Ε, είναι πραγματικά επέσχυντη αυτή η μεταφορά, χιλιάδε χιλιόμετρα ε, σε συνθήκε τρομερή ζέστη, κάψωνα και πάει αυτό σε εργοστάσια αλαντικών και φτιάχνουν σαλάμι στην Νότια Ιταλία από άλογα χρειάζεται πραγματικά βελτίωση, ειδικά για τους ύπους, είναι τραγικές οι συνθήκες. Ε, κύριε Επιτροπή, κατανοώ ότι μόλις αναλάβατε, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ε, αυτή η επιστημονική δουλειά έχει ήδη γίνει. Αυτό που προτείνεται για το 8ωρο έχει ήδη μελετηθεί. Για τα υποειδή είπαμε, υπάρχει αυτή η μελέτη, την έχετε και σας παρακαλώ να το χρησιμοποιήσετε και να το χειριστείτε ως προτεραιότητα. Υπάρχουν τα επιστημονικά στοιχεία και παρακαλώ να είναι ε, η πρώτη ε, προσέγγιση για ένα κανονισμό πεφωτισμένο για τη μεταφορά των ζώων. Ευχαριστώ κύριος Γκούσταυσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι ε, στον κόσμο μας ε, σήμερα να αποσυνδέονται τόσο πολύ από τη φύση, να αλωτριώνονται και να μην σέβονται τα άλλα είδη ε, ζώων των οργανισμό. Υποφέρουν τα ζώα τα μεταφέρονται σε τόσο μεγάλες αποστάσεις. Και είναι πραγματικά πολύ μικρά τα οχήματα αν δεν τηρήσουμε το οκτάωρο, για προσπαθείτε να ταξιδέψετε με 8 αγελάδες σε ένα δίκλινο κρεβάτι μέσα σε ένα ε, φορτηγό. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να ζητούμε ανέφικτα πράγματα, αλλά ε, αυτό το ζήτημα της μέγιστης διάρκειας 8 ωρών ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί και είναι και, πολύ μεγάλο το οκτάωρο ως διάστημα. Και δεν θα πρέπει τα χρήματα να είναι πιο σημαντικά από τη ζωή την ίδια. Η κυρία Ράντς Γκαρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εγώ είμαι κατά της θέσπισης νέων κανόνων για την ευζοία, όταν ο ισχύων κανονισμός ήδη προβλέπει διατάξεις που ρυθμίζουν τη διάρκεια του ταξιδιού ανάλογα με το είδος του ζώου και με βάση τις επιστημονικές γνώσεις που διαθέτουμε. Μην ξεχνάτε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων, η ΕΦΣΑ, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει επιστημονική βάση που να τεκμηριώνει την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Και η ευημερία των ζώων, η ευζοία, εξαρτάται από την ποιότητα του ταξιδιού, από τις συνθήκες του ταξιδιού, από τη μεταχείριση των ζώων και από τον κατάλληλο εξοπλισμό των οχημάτων. Μην ξεχνάτε ότι οι μεταφορείς ε, ήδη υποχρεούνται να τηρήσουν κάποιες προδιαγραφές, ελάχιστη πυκνότητα, εξαρισμός, θερμοκρασία, ε, διάρκεια ποτίσματος, ε, τροφή, παροχή τροφής. Και νομίζω ότι η σωστή εφαρμογή τη κοινοτική νομοθεσία είναι υπεραρκετή για την εξασφάλιση τη ευζοία στη μεταφορά. Το πρόβλημα είναι ο χαμηλό ρυθμό και βαθμό συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν του ελέγχου και τι επιθεωρήσει για να εξασφαλίσουμε συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία. Αντί να εισάγουμε περιορισμού στην ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων που δεν θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα σε όλε τι χώρε και θα ευνοήσουν ορισμένα εμπορικά συμφέροντα ει βάρο άλλων αν είναι αλήθεια ότι βασανίζονται στα μακροχρόνια ταξίδια, μα, μακρόρα ταξίδια, τότε να μην περιορίσουμε την ομοθεσία αυτή μόνο στα ζώα φαγή, να τα εκτείνουμε και στη μεταφορά ζώων προ πάχυνση. Γιατί αυτέ οι διακρίσει. Όλα τα ζώα έχουν δικαίωμα σε αξιοπρεπή μεταχείριση και πιστεύω ότι στην περίοδο αυτή τη οικονομική κρίση που διανύουμε δεν είναι η καταλληλότερη στιγμή για να υποβάλουμε νέε προτάσει που δεν ε, θεμελιώνονται καν επιστημονικά. Δεν ε, είναι σωστό να υποβάλουμε τέτοιου είδους ρυθμίσει. Ευχαριστώ κύριε Σολέιντσακ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να υποστηρίξω την πρωτοβουλία αυτή και την έκθεση και να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας Βοητσεχόφσκι για, την, για το διαλεκτικό του πνεύμα, για την αναζήτηση συμβαστικών ε, τροπολογιών και συμφωνιών και με συνεχές μέλημα την ευζοία. Το 2005 εγκρίθηκε ο σχετικός κανονισμός και ε, τότε θυμάμαι ότι πολλοί διαρωτήθηκαν αν αξίζει μια τέτοια νομοθεσία. Σήμερα όμως οι μελέτες και η εμπειρία μας δείχνουν ότι ο κανονισμός ήταν ένα πολύ καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι το βήμα αυτό έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βελτιώθηκε η ευζοία, η καλή διαβίωση των ζώων και βελτιώθηκαν και οι οικονομικές συνθήκες και για τους γεωργούς κτηνοτρόφου αλλά και για τους επιχειρηματίες. Και αυτό είναι σήμερα ε, το, το μέτρο που μας δείχνει ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι. Ο περιορισμό τη μέγιστη διάρκεια μεταφορά είναι πολύ καλή και συνετή πρόταση. Πολύ λογική. Γιατί έτσι θα ενισχύσουμε την τοπική παραγωγή, τα τοπικά σφαγεία, θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης ε, στις τοπικές κοινότητες, εκεί που περισσότερο ε, χρειάζονται αυτές οι θέσεις. Και άλλωστε θα περιορίσουμε και το κόστος, κάτι που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η μεταφορά των ζώων σε μεγάλες αποστάσεις αυξάνει το κόστος και ένα τμήμα του κόστους με επιβαρύνει τους καταναλωτές γιατί τα προϊόντα είναι ακριβότερα από ό,τι θα έπρεπε κανονικά να είναι. Επίσης είναι σημαντικό το ότι σήμερα παρά τις διατάξεις και περί αυτού πρόκειται και το επισημαίνουμε αυτό στην έκθεση ε, και απευθύνουμε έκθεση στα κράτη-μέλη για τις κτηνιατρικούς ελέγχους. Παρά τις διατάξεις, οι διαδικασίες που ε, υπάρχουν στα χαρτιά δεν τηρούνται πιστά. Ε, όχι μόνο για τη μεταφορά, αλλά και για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των ζώων. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ε, πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό προκειμένου να βελτιωθεί η ευζοία. Σας ευχαριστώ. Πρίτα Ράιμαρτ, επόμενη συνάδελφος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, στο θέμα της μεταφοράς των ζώων ε, τα συναισθήματα χτυπάνε κόκκινο γιατί βλέπουμε εικόνες ε, ζώων που μεταφέρονται που δεν είναι απαραίτητα αυτό που θα θέλαμε να δούμε. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα υπάρχουν διατάξεις, κανονισμοί που δεν εφαρμόζονται και ούτε και διεξάγονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις εικόνες. Όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι οδηγίες και οι κανονισμοί πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν τα αίτια του γιατί έχουμε μακρινές αποστάσεις στην Ευρώπη. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε θεσπίσει τις διατάξεις, ε, ε, προβλέπουμε υψηλότερες υγιεινές προδιαγραφές ε, καλύτερους ελέγχους υγείας. Ε, βέβαια με τον τρόπο αυτό χάσαμε πολλά σφαγεία που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο κόστος. Αν θέλουμε μικρότερες αποστάσεις πρέπει να αλλάξουμε τις ε, συνθήκες πλαίσιο και εν πάση περιπτώσει αυτή η οδηγία για την προστασία των ζώων εφαρμόζεται σε όλα τα κρατημέλη και να διεξάγονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το εξής εφόσον ε, έχουμε μικρές ε, αποστάσεις ή ε, πολλοί βγαίνουν από τον ανταγωνισμό, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πιστεύω λοιπόν ότι η έκθεση που κατέθεσε ο κύριος Ουτσέφσκι είναι πολύ καλή και θα τη στηρίξουμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Ε, συνάλφος Σμιθ Άλλαν. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ε, θα ευχαριστώ επίσης, ε, θα συγχαρώ ε, τον εισηγητή, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, κατέληξε σε ένα λειτουργικό συμβασμό σε αυτά το συναισθηματικά φορτισμένο θέμα σας καλωσορίζουμε ε, σε αυτή την ε, πρώτη σας συζήτηση. Ελπίζουμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Ε, εμείς θέλουμε να αποφύγουμε τη βιότητα κατά των ζώων και θα συμφωνήσετε ότι το πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε με αυτή την έκθεση είναι να κάνουμε απολογισμό που βρισκόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους κανόνες, να τους εφαρμόζουμε πρέπει αυτούς που υπάρχουν. Ε, οι, αιτία, πολλές φορές λέμε, δεν έχει αποδειχθεί ότι πρέπει να υπάρξουν ε, νέες διατάξεις. Αυτό ε, δεν στηρίζεται και από την επιστήμη. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για μικρά σφαγεία. Είπατε ε, ότι διαφωνείτε στο να υπάρχει μεγαλύτερο κόστος. Δύσκολα τα οικονομικά, αλλά θέλω να σας μεταφέρω κάποιες πληροφορίες από την Σκοτία, όπου έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αν ακολουθήσουμε την αντίθετη κατεύθυνση αυτό θα είναι αρνητικό. Θέλω να συνεργαστώ μαζί για να καταλήξουμε σε πιο θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριο Πέτερ Βαντάλεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο Βοητσεχόφσκι, εξαιρετική του η έκθεση και καλωσορίζουμε τον νέο επίτροπο. είμαι υπέρ της πρότασης ε, της μέγιστης διάρκειας 8 ώρων για τα ζώα προς ε, σφαγή. Θα πρέπει να είναι πιο αξιοπρεπής οι συνθήκες. Θα πρέπει να δούμε όμως ε, πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη μεταφορά σφαγίων, δηλαδή σφαγμένων ζώων και όχι ζώων προς σφαγή. Καλύτερα τρώω εγώ ένα κρέας που έχει μεταφερθεί πολλές ώρες παρά ένα κρέας από ζώο που έχει μεταφερθεί πολλές ώρες και έχει στρεσαριστεί. Σε πολλές χώρες βλέπουμε ότι υπάρχει υπερβολική ε, κριτική ε, για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι επιθεωρήσεις ή κρεοσκοπικοί έλεγχοι και στα σφαγεία ε, και αυτό θα πρέπει ε, να κοιτάξουμε τους ελέγχους και να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ζώων αλλά και τη μεταφορά των κρεάτων. Παρακαλώ τον Επίτροπο να εργαστεί και εκεί. Ε, ο κύριος Κλάτφελτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ κανονικά είμαι κατά των νέων μέτρων για την προστασία των ζώων γιατί έτσι υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα ε, γιατί συχνά έχουμε ανταγωνιστές ε, που δεν ε, τηρούν τις ίδιες προδιαγραφές με εμά και μεταφορές από μεγαλύτερες αποστάσεις σημαίνουν και μεγαλύτερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό το θέμα λοιπόν σε εθελοντική βάση, αλλά υποστηρίζω το ζήτημα της μέγιστης διάρκειας μεταφορών 8 ωρών δεν αφορά μόνο την ευημερία των ζώων, αφορά και την οικονομία ε, λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, άρα και καλύτερη κατάσταση του κλίματος. Λόγω αυτού του περιορισμού λοιπόν των 8 ωρών, δεν μπορούν να έρχονται ζώντα ζώα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε να πηγαίνουν εκεί και να σφάζονται με συνθήκες εκτρές. Ε, εμείς έχουμε πολύ καλύτερες συνθήκες ε, στα σφαγεία μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μην αφήνουμε παραθυράκια στο σύστημα και να μην επιτρέπονται εξαιρέσεις και στρεβλώσεις και να μην μπορεί κανείς να παρακάμπτει αυτή τη μέγιστη διάρκεια μεταφοράς οκτώρων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προωθηθούν τα μικρά σφαγεία, ε, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και στις περιφέρειες ε, στην Ήπεθρο. Γι' αυτό υποστηρίζω αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεκάστρο. Presidente, caro Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον ε, εφαρμογή του κανονισμού του 2005 για την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αποκαλύπτει ότι στα κράτη-μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Και θέλω να επενθυμίσω ότι αυτή η νομοθεσία είναι η πιο προχωρημένη σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Επιτροπή Γεωργίας, την οποία εκπροσωπώ, πρόσεξε πάρα πολύ καλά το όλο θέμα, ισόρροπη η και ε, στην έκθεση Επιτροπής έχουμε εντοπίσει κάποια κενά σχετικά με τα ε, στοιχεία και κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη να περιστούν οι ώρες για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή αυτό είναι σημαντικό αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άκαμπτες υγειονομικές διατάξεις που έχουμε επιβάλει δεν μπορούν να εφαρμοστούν πολλές φορές από τα μικρά σφαγεία δεν μπορούμε βέβαια να περιορίσουμε την συζήτηση και να πλουστεύσουμε να, πούμε, να μιλάμε μόνο για ώρες υπάρχουν και άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την καλή διαβίωση των ζώων παραδείγματος χάρη να είναι σωστή υποδομή του οχήματος, ε, να έχουν τοποθετηθεί σωστά τα ζώα, όπως έχει υποδειχθεί και από την ΕΦΣΑ. Ευχαριστώ τον εισηγητή Βατσεβόσκη και τους σκιώδης εισηγητές για τη θαυμάσια δουλειά που έχουν κάνει και τους καλώ να υπερψηφίσουν την έκθεση που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από την Επιτροπή Γεωργίας. Ο κύριος Τσανόνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, 1.100.000 πολίτες μας ζητούν να περιορίσουμε σε 8 ώρες ε, την ε, μεταφορά των ζώων που πάνε για σφαγή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να είναι άκαμπτο μπροστά σε ένα τέτοιο αίτημα πολιτισμού. Αν θέλουμε να προστατεύουμε τα ζώα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους πρέπει να πούμε φτάνει πια με αυτά τα ε, ταξίδια μια ολόκληρη μέρα ε, που κάνουν τα ζώα να υποφέρουν πάρα πολύ. Ε, κύριε Επίτροπε, ο κανονισμό δεν επιτρέπει αποτελεσματικού ελέγχου σε μακρέ ε, διαδρομές και συμβαίνει συχνά τα ζώα να μεταφέρονται με ε, τραγικές συνθήκες χωρίς εξαρισμό, με πολύ λίγο νερό, ε, σε πολύ μικρό χώρο. Να ψηφίσουμε λοιπόν για τις 8 ώρες όπως αναφέρεται και στην γραπτή δήλωση του Μαρτίου αυτού του έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να είναι ειδοποιός διαφορά γιατί με αυτή την ε, ψηφοφορία έχουμε επιτέλους δυνατότητα να θέσουμε τις βάσεις για να μην υποφεύγουμε περιτά εκατομμύρια ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριο Σεκέρσκι. Ευχαριστώ. Ούτε και εγώ είμαι υπέρ τη μέγιστη μεταφορά. Αναφέρθηκε ο περιορισμό στι 8 ώρε. Εγώ θα προτιμούσα να είναι 6 ώρε η μέγιστη διάρκεια μεταφορά των ζωντανών ζώων. Γιατί το θέμα του περιορισμού τη μεταφορά είναι πολύ δυσχερέ πρόβλημα. Γιατί καλό είναι να ενισχύσουμε τα τοπικά σφαγεία που ε, μπορούν να αυξήσουν τη, το δυναμικό τους, τη δραστηριότητά τους και αυτό αποβαίνει και προς όφελος ε, του περιβάλλοντος ε, και έτσι θα περιοριστούν οι μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε και τις συνθήκες μεταφοράς, εξαρισμό, ποτίστρες και σωστή κατάρτιση των μεταφορέων. Μεγάλες μεταφορές επιβαρύνουν ιδιαίτερα και τους καταναλωτές ε, και βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διασυνοριακές μεταφορές ε, και εκεί υπάρχουν προβλήματα γιατί οι περιορισμοί στην, στη διάρκεια μεταφοράς θα τονίσει ε, τις τοπικές διαφορές αλλά δεν θα πρέπει να εμποδίσουμε τη δυνατότητα εξαγωγών των διαφόρων παραγωγών. Ε, είναι σημαντικό να τηρηθούν οι προδιαγραφές ε, για την φόρτωση-εκφόρτωση, για τις περιόδους ε, ανάπαυσης και να αποφευθεί όσο γίνεται το στρες των ζώων. Επίσης, να μην τραυματίζονται χωρίς λόγο ή να μην επιδεινώνονται οι συνθήκες ασφαλείας τους με τις νέες διατάξει για τις μεταφορά στι μεγάλε αποστάσει θα πρέπει να, να καταλήξουμε σε μια συνετή και ορθολογική απαραίτητη λύση. Γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ε, ευζοία, την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά και το περιβάλλον. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες μεταφοράς και συμφωνώ με τον εισηγητή. Και μήπως ήταν πιο ανθρωπιστικό, να δώσουμε μια άλλη λύση για τα ζώα. Ευχαριστώ κύριος Γιώργενσεν. Κύριε Επίτροπε, εγώ είμαι γενικά ευγενής, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι αυτό που επιδείξατε εδώ προηγουμένως είναι αλαζονία και καθόλου δημοκρατικό να λέτε σε ένα εκατομμύριο πολιτών που ζήτησαν περιορισμό της διάρκειας μεταφορών ότι παραμένετε αδιάφορος απέναντι ε, σε αυτό το αίτημα. Γιατί δεν υπάρχουν, λέει, επιστημονικά δεδομένα. Μα το Κοινοβούλιο σε γραπτή του δήλωση δέχτηκε να ζητήσουμε τροποποίηση των κανόνων για τη διάρκεια της μεταφοράς. Δεν μπορείτε να λέτε ότι παραμένετε αδιάφορος. Επαναλαμβάνω, είναι αλαζονία αυτό. Ε, για τα επιστημονικά δεδομένα. Λες και δεν υπάρχουν στοιχεία. Θα μπορούσαμε να πούμε ε, η μέγιστη διάρκεια μεταφοράς όλων των ζώνων είναι 8 ώρες. Οι Ευρωπαίοι κτηνίατροι δεν είναι επιστήμονες. Είναι συναισθηματική η προσέγγιση του και ε, παρακαλώ να είστε πιο σωστός απέναντι στους πολίτες. Η κυρία Κιώστιγκερ, ευχαριστώ. Πρόεδρε, με την έκθεση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, βοηθάει ε, για τη μεταφορά των ζώων. Είναι κυρίως εθνική αρμοδιότητα αυτό και τα κράτη-μέλη ε, με διαφορετικό τρόπο τα προσεγγίζουν. Και από πολλές ε, πλευρές ε, χρειάζεται ρύθμιση. Δεν υπάρχει περιορισμό σε πολλές χώρες και τα εγωπρόβατα και τα βοηδή μπορεί να μεταφέρονται μέχρι και 29 ώρες μέχρι το σφαγείο. Ταυτόχρονα επίσης θα πρέπει να δούμε αλλιώς από άλλη πλευρά το ερώτημα. Δυστυχώς ε, έχουν ε, υπάρξει ρυθμίσεις για τα σφαγεία που οδήγησαν στο κλείσιμο πολλά τοπικά και περιφερειακά σφαγεία. Θα πρέπει τα ζώα να σφάζονται όσο γίνεται πιο κοντά στον τόπο εκτροφής τους. Και βέβαια θα πρέπει ε, να ξέρουμε ότι υπάρχουν ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, ορεινές που είναι δύσκολη στην πρόσβαση. Αλλά αυτό που έχει σημασία για την προστασία των ζώων δεν είναι μόνο η διάρκεια αλλά και η ποιότητα της μεταφοράς. Θα πρέπει να είναι οι προδιαγραφές ε, ε, οι πιο σύγχρονες ε, για τα φορτηγά, για τη φόρτωση, θέματα ποτίσματος, ταΐσματος και εξαρισμού να γίνονται σεβαστά. Επίσης οι προδιαγραφές περίπου εναρμονισμένες είναι και ένα θέμα ανταγωνισμού και τελικά εξυπηρετούν και τους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Η κυρία Ουλρίκε Ρόντος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι και εγώ υπογράψαμε την ε, δήλωση αυτή. Δηλαδή να περιστεί η μεταφορά των ζώων προσφαγή σε 8 ώρε. Γιατί όσο μακραίνει η διαδρομή υποφέρουν πιο πολύ τα ζώα. Και δεν είναι απαραίτητο τα ζώα προσφαγή. Γενικά τα ζώα να τα μεταφέρουμε περισσότερο από 8 Πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να περιοριστούν οι διαδρομές. Όπως και οι συνθήκες ε, των μεταφορών είναι καθοριστικές. Το αίτημα ε, να υπάρχουν εξαιρέσεις ε, λόγω ε, κυκλοφοριακής συμφόρησης ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων, αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Άλλο τώρα το θέμα των απομακρυσμένων περιοχών λόγω των υγιεινών προδιαγραφών ε, πολλά μικρά σφαγεία έκλεισαν. Αυτό έπρεπε να το εμποδίσουμε. Παρότι πρέπει να πω οι προδιαγραφές ε, είναι καλές αλλά έπρεπε να βοηθήσουμε τα μικρά σφαγεία. Ε, να γίνουν πιο οικονομικά, πιο αποδοτικά τα μικρά σφαγεία, αυτό το στηρίζω. Και με τον τρόπο αυτό με, δυο, με ένα σμπάρο, δυο τριγώνια. Γιατί μπορούμε να αποφύγουμε τις ε, μεγάλες διαδρομές, να δημιουργήσουμε υπεραξία επιτόπου και επίσης και θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ κυρία Πατράων Νέβες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μα και του και εισηγητέ για τι άκουνε προσπάθειε του και την αναζήτηση ισορροπημένη λύση μεταξύ των αντικρώμενων συμφερόντων, Αφενό των ε, ζώων, της ευζοίας, της καλής διαβίωσής τους, αλλά και των ανθρώπων ε, που θα πρέπει να βελτιώνουν το βιωτικό τους επίπεδο, όχι όμως βάρος των ζώων. Επίσης, μεταξύ των εκτροφέων, των κτηνοτρόφων, των παραγωγών δηλαδή ζώων, και της ανάγκης ε, προσοδοφόρας δραστηριότητας βρέθηκε μια σωστή ισορροπία. Ε, βέβαια, η μέγιστη διάρκεια των οκτώρων δημιουργεί προβλήματα στις περιφερειακές χώρες ε, όπως η Πορτογαλία. Γιατί με υποχρεωτικές πολλές ε, διακοπές στο ταξίδι και τη μέγιστη διάρκεια δημιουργούν, δημιουργείται τεράστιο κόστος, μεγάλο άχθος και έρχεται σε ε, δυσμενή μεταχείριση το, το απομακρυ... περιφερειακό κράτος ή εξόχως απόκεντρη περιοχή. Δεν μπορεί να ισχύει η μέγιστη διάρκεια των 8 για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές όπως ενέκρινε η Επιτροπή ε, Γεωργίας. Γιατί κάτι τέτοιο θα απέτρεπε, ουσιαστικά θα απαγόρευε την εξαγωγή ε, ζώων, τη μεταφορά ζώων από τις εξόχως απόκεντρε περιοχές προς την υπηρετική Ευρώπη. Οι εξόχως απόκεντρε περιοχές είναι ήδη σε μειονεκτική θέση εξαιτία τη γεωγραφική του ε, θέση και δεν μπορούμε να επιδεινώσουμε την κατάστασή τους ε, επιβάλλοντας περαιτέρω περιορισμούς που τους πλήττουν εξαιτία τη γεωγραφική του θέση ουσιαστικά. Ευχαριστώ κύριο Σάλβε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η προστασία των ζώων και της ευζοίας τους αποτελεί πολιτιστικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινωνία της. Φυσικά θα πρέπει εμείς πολιτικοί να μετατρέψουμε σε προσανατολισμούς το, το αίσθημα του πολίτη Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε σωστές συνθήκες μεταφοράς για τα ζωντανά ζώα, με προδιαγραφές και επιστοποίηση των οχημάτων, με ε, κατάλληλους ε, ελέγχους και επιθεωρήσεις, τους παραγωγούς, οργανωτές, ε, μεταφορές, σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές αρχές και με τους προσανατολισμούς που έχουμε καθορίσει. Βέβαια, και εφόσον συντρέξουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τα επιστημονικά πορίσματα και να λάβουμε υπόψη κάποιες ε, προϋποθέσεις, ε, κυρίως γεωγραφικές, κυρίως των περιφερειακών και εξόχων απόκεντρων περιοχών, που δεν συνάδουν με την εισαγωγή της ε, μέγιστης διάρκειας σε 8 ώρες. Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την κοινή λογική ώστε να κρίνει ότι σε ορισμένε περιπτώσει ο περιορισμό τη μέγιστη διάρκεια 8 ώρε είναι ανέφικτο. Και μετά του ομιλητέ που ήταν εγγεγραμμένοι για τη συζήτηση, ακολουθεί το σύστημα Κατσία ή το λόγο έχει η κυρία Μαγκίνε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και όλους τους σκιώδεις που εργάστηκαν σε αυτή τη δύσκολη πλήν όμως σημαντική έκθεση. Ε, θα ήθελα να ευσύσω την προσοχή σας στην πρώτη παράγραφο και συνοψίζει όλες τις ανησυχίες και τονίζει ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζεται σωστά η ισχύουσα νομοθεσία και οι νόμοι στα κράτη-μέλη. Ε, δεν χρειάζεται να ζητήσουμε περισσότερη νομοθεσία. Αν δεν εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες, τι νόημα έχει να βάλουμε επιπλέον ένα στρώμα κανόνων αφού υπάρχουν ήδη προβλήματα. Επίσης, σε αυτό τον καιρό της λιτότητας αναρωτηθώ αν τα κράτη-μέλη θα μειώσουν τους πόρους για τις επιθεωρήσεις ε, στη μεταφορά των ζώων. Γιατί ακριβώ δεν έχουν τα χρήματα για να τους υλοποιούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξει πολύ προσεκτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα δεύτερο θέμα και το ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι είναι το θέμα της συγκέντρωσης των σφαγείων ε, με ΕΙ. Το είπε και η κυρία Γέγλε και οι υπόλοιποι. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι συμβαίνει αυτό σε σχέση με τη συγκέντρωση. Όχι μόνο για την ευημερία των ζώων, αλλά και για την ε, υπόθεση του ανταγωνισμού των παραγωγών. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. πάρα πολύ σοβαρό. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας στήσω την υπερψήφιση της έκθεσης ε, ε του κ. Βοτσεχόφσκη που προτείνει περιορισμό της μέγιστης διάρκειας ε, των ζωντανών ζώων προσφαγής 8 ώρες. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται και πολύ σημαντικές ε, τρεις τροπολογίες που μιλούν για τη βελτίωση των συνθήκων μεταφοράς και την ε, διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων. Εδώ και πολύ καιρό, και εδώ θα ήθελα να ε, αποδείξω γιατί είναι σημαντική και θα πρέπει να υποστηριχθεί η μέγιστη διάρκεια σε 8 ώρες, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, δεν ε, λαμβάνει υπόψη πολλές επιστημονικές μελέτες που μιλούν για την ανάγκη τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και τη θέσπιση περιορισμού της μέγιστης διάρκειας 8 ώρες. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ευρεία συζήτηση για το θέμα αυτό και να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού τη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις ζωντανών ζώων για σφαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Now I'll give the floor to colleague ε, Richard Howitt. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Richard Howitt. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ε, εξ ονόματος ε, της μη κυβερνητικής οργάνωσης που αφορά την ευημερία των ύπων και εδρεύει στην εκλογική μου περιφέρεια, θα ήθελα να πω ότι μας απαντήσατε πρόεδρε, αλλά δεν είπατε ότι 65.000 άλογα μεταφέρονται σε μακρές αποστάσεις κάθε χρόνο, διανύουν την Ευρώπη ολόκληρη και 94% έχουν ε, μια αοξία πληγή, 90% εμφανίζουν συμπτώματα ασθένειας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λέγει ότι χρειάζεται καλύτερη εφαρμογή αλλά το ψήφισμα λέει ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπάρχουν αρκετές εφαρμογές αν δεν είναι σωστοί οι κανόνες από την αρχή τους. Υπάρχουν ευρήματα ε, επίσης και του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων και άλλα επιστημονικά. Την περασμένη ε, Παρασκευή ε, ε, είδα στην εκλογική μου περιφέρεια να στέλνουν 4.500 κάρτες στον πρόεδρο Μπαρόσο για να σταματήσει αυτή η μεταφορά λόγων προς την Ιταλία. Χαίρομαι ε, που δίνει μια δεύτερη ευκαιρία για τα τραυματισμένα ε, άλογα αυτή η οργάνωση. Ε, θα ήθελα να μπορώ να είμαι και περήφανος για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε λιγότερα άλογα να σώσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Χόιτ. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κύριος Νικουλέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες συμμερίζονται τις ανησυχίες μας και προβληματίζονται για τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων. Ένα θέμα συναισθηματικά φορτισμένο και προκαλεί σποδρές συζητήσεις. Οι απάνθρωπες συνθήκες μεταφοράς είναι απαράδεκτες. Θα πρέπει να τις βελτιώσουμε. Όλοι θέλουμε κάτι τέτοιο. Αλλά περισσότερο με αυτό να ασχοληθούμε με την ε, εισαγωγή σωστών συνθηκών μεταφορά και όχι με τον περιορισμό τη μέγιστη διάρκεια του ταξιδιού. Έχουμε πολλού κανόνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εφαρμόζονται λοιπώς όμω. Ούτω ή άλλω ε, τα ζώα υποφέρουν. Μιλήσαμε για την επαναφορά των τοπικών μικρών σφαγείων. Αυτό είναι σημαντικό και θα περιορίσει τι μεταφορέ σε μεγάλε αποστάσει. Ελπίζω η μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική να το λάβει υπόψη. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή είναι ο συνάδελφο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή μας. Η Σλοβενία είναι μια χώρα διαμετακόμισης Οπότε, με βάση την προσωπική μου εμπειρία, θεωρώ ότι όντω υπάρχει πρόβλημα στη μεταφορά των ζώων εξαιτία κακών συνθήκων. Ήμουν μάρτυρα μια τέτοια κατάσταση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί βέβαια και η εφαρμογή του κανονισμού 1 του 2005. Είμαι υπέρ και τη μέγιστη διάρκεια 8 ώρε. Το σύστημα όμω θα πρέπει να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και να είναι τέτοιο που να δίνει ενάψματα για καλύτερη μεταχείριση των ζώων. Είναι κρίμα να βασανίζουμε τα ζώα που προορίζονται για σφαγή. Άλλωστε, το στρες αυτό επηρεάζει και την ποιότητα του κρέατος. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ζώα ταξιδεύουν στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Έχει διπλασιαστεί ο αριθμός τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει εσωτερική ενιαία αγορά. Τίθεται και θέμα κέρδους αλλά πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και στις ιδιαιτερότητες, στη διαφορετικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και, ε, και να δώσουμε έμφαση στην τοπική παραγωγή και κατανάλωση. Ευχαριστώ. Πολύ κύριε Σβέρ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κοφεράτη. Grazie Presidente. Signor... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όπως αναφέρθηκε ήδη, η έκθεση της Επιτροπής ε, είναι μια ένδειξη πολιτισμού, ε, κυρίως στους κανόνες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά όλα σε σχέση με το θέμα που συζητάμε. Μιλάμε για ανθρώπινα όντα, για όντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την υγεία μας. Και τρία πράγματα είναι απαραίτητα. Το πρώτο είναι η εισαγωγή μιας αυστηρής δέσμης δέσμευση των 8 ώρων κατά το μέγιστο για τη μεταφορά. Δεύτερο, συνθήκες μεταφοράς, ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται τα ζώα αυτά από το ένα σημείο στο άλλο δεν ε, είναι σημαντικό ε, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι οι συνθήκες ε, γιατί εμείς τελικά θα χρησιμοποιήσουμε το κρέας τους και τέλος νομίζω ότι ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλεγχη πάρα πολλές φορές οι συνθήκες που ορίζουμε εμείς παρακάπτονται, παραμβιάζονται είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχουν έλεγχοι και κυρώσεις γιατί ένας κανόνας που εφόσον έχει αποφασιστεί πρέπει και να εφαρμόζεται Τελευταία ομιλήτρια, η συνάδελφος κυρία Κάντενμπαχ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, ευχαριστώ που έχω και πάλι την ευκαιρία να μιλήσω, ε, διότι επειδή με κατέκλυσαν τα συναισθήματα προηγουμένως που μίλησα εξ ονόματος της ομάδας μου, ξέχασα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή συνεργασία. Ακριβώς είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένο το θέμα και κατάφερε ωστόσο να έχει ένα ισορροπημένο κείμενο στην έκθεσή του και πραγματικά να προστατεύει τα ζώα με το σωστό τρόπο. Θα ήθελα παραμονές Χριστουγέννων, μια που μιλάμε για την προστασία των ζώων, να μην λησμονήσω να πω ότι τα ζώα είναι ζωντανά πλάσματα, έχουν δικαίωμα στην προστασία και δεν είναι αντικείμενα ε, για δώρα. Δηλαδή, όσοι θέλουν να χαρίσουν δώρο σε κάποιον σκεφτούν και τα ζώα, ε, αυτά που περιμένουν ε, στα κοινοκομεία να βρουν μια οικογένεια. On behalf of the της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο κύριο Τόνιο Μπόρτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην πρωτομιλία μου ξεκαθάρισα ότι δεν ήμουν ικανοποιημένο με τον τρόπο που εφαρμόζει το κανονισμός. Δεν προσπάθησα να αποφύγω την απάντηση. Ενημέρωσα το Κοινοβούλιο για τα μέτρα που θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν. Στο βαθμό που υπήρχαν διαδικασίες επί παραβάση, έχουν αρχίσει και έχουν υπάρξει και 14 ε, ανακοινώσει επικοινωνία με τα κράτη-μέλη και δύο εκκρεμούν ακόμα. Συμμερίζομαι όμω την άποψη εκείνων που λέγουν ότι αν δεν είμαστε καν σε θέση να εφαρμόσουμε τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις, πόσο δυσκολότερο θα είναι να εφαρμόσουμε νέους κανόνες και νέα νομοθεσία. Ήμουν σαφέστατος στην εξήγησή μου ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προτείνει νέα νομοθεσία αλλά καλύτερη εφαρμογή της συγκεκριμένης. Εγώ μπορώ να σας υποσχεθώ μόνο αυτό που μπορεί κατά τη γνώμη μου να ε, κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας επισήμενα τους τομείς που γίνεται αυτό ως προς την εφαρμογή και τι θα ενισχυθεί. Πρώτον, να εναρμονιστούν οι αναφορές των κρατών μελών σχετικά με τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, γιατί ούτε αυτό δεν έχουμε. Δεν έχουμε μια ενιαία ε, μορφή ε, αναφοράς για την υλοποίηση και επιβολή του κανονισμού του 2005. Θα διεξαχθεί επίσης και διάσκεψη στο Δουβλίνο το 2013 για αυτό το ειδικό θέμα και για τη μεταφορά των ζών. και το 2013 επίσης θα ε, ξεκινήσει μια νέα σειρά μελετών και επισκέψεων επιτόπου και θα συμμετέχουν όχι μόνο τα κράτη-μέλη αλλά και ένας ελεγκτής, ένας επιθεωρητής από το FVO, το Γραφείο Τροφίμων και Εκτινιατρικών Θεμάτων. Και θα καθοδηγεί καθώς και θα συνοδεύει επιθεωρητές και ελεγκτές ε, των κρατών μελών και θα ακολουθεί και τις παραδοσιακές οδούς μεταφοράς ζώων. Επίσης θα βελτιώσουμε του ελέγχου στη μεταφορά των ζώων καλύτερα, με καλύτερη χρήση συστημάτων πλοήγησης. Γιατί υπήρχαν κύριε Πρόεδρε μεγάλα προβλήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή όμω έχουμε τη, στη διάθεσή μα αυτή τη σύγχρονη τεχνολογία που δεν είναι και πολύ δαπανηρή. Θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε καλύτερα. Αυτό σήμερα δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχει ούτε εναρμόνιση ούτε η βούληση εκείνων που ενέχονται σε αυτά τα θέματα για να έχουν τα συστήματα πλοήγηση θα το κοιτάξουμε με τις νομικές υπηρεσίες να φροντίσουμε να δούμε αν υπάρξει ε, χώρος να εισαχθεί με τρόπο υποχρεωτικό και δεσμευτικό. Ε, αυτή λοιπόν είναι η εισαγωγική μου τοποθέτησή σήμερα. Αλλά δεν είναι η τελική προσπάθεια. Η αρχή είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας και του κανονισμού. Κάτι που μπορεί να είναι και λογικό και φιλόδοξο. Αν αποτύχουν τα πάντα και η εφαρμογή, αν δεν λειτουργήσει σωστά, που πιστεύω ότι θα λειτουργήσει, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη θέση μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, δίνω τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Γιάννους Βοτσεχόφσκι, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους ε, ευρωβουλευτές που έλαβαν το λόγο και συμμετείχαν στη συζήτηση. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις τους και ε, εκείνες που ήταν υπέρ της έκθεσης και ε, τους συναδέλφους που άσκησαν επικρίσεις. Πάντως ήταν αγαστή συνεργασία με τους συναδέλφους και τους ευχαριστώ θερμά γιατί ήταν δύσκολη έκθεση ε, δεν φανταζόμουν όταν ανέλαβα την έκθεση αυτή ότι θα ήταν μια έκθεση τόσο συναισθηματικά φορτισμένη που θα προκαλούσε τόσο έντονα συναισθήματα και πάθος στη συζήτηση. Η έκθεσή μου ε, είναι καρπός συμβιβασμού. Είχαμε αφενός ε, πολύ αυστηρές προτάσεις για περιορισμό της μέγιστης διάρκειας, ε, είχαμε από την άλλη πιο χαλαρέ προτάσει για να μην ασχοληθούμε καθόλου με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι ο συμβασμό στον οποίο κατέληξα είναι πολύ συνετό και λογικό και σα παρακαλώ να τον υποστηρίξουμε στην αυριανή ψηφοφορία. Αύριο ε, έχουμε 12 δωδεκάτου του 2012 και στις 12 το μεσημέρι θα ψηφίσουμε. Ελπίζω λοιπόν αυτό το 12 που εμφανίζεται τόσες πολλές φορές να είναι γούρικο για την έκθεσή μου και να υπερψηφιστεί. Ε, και πιστεύω ότι χάρη σε αυτήν θα συμβάλλουμε στη βελτίωση των συνθήκων μεταφορά των ζωντανών ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για μια ακόμη φορά σα ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο συγητή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίσω περιομένη την συζήτηση. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.30. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και αφορά στη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Πρόκειται για προφορική ερώτηση Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Ε, δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στη συνάδελφο κυρία Αρλέν Μακάρθη, που είναι συντάκτης για πέντε λεπτά. The floor is yours. Thank you. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι έχουμε τη